κάνω ε, μία ανακοίνωση. Λάβαμε στις ε, υποψηφιότητες του ECR για τις ε, επιτροπές, τις διακοινοβουλευτικές επιτροπές υπάρχουν στα πρακτικά και αν δεν υπάρχουν ενστάσεις θα θεωρηθούν εγκεκριμένες αυτές.